Pan Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακαλώ λάβετε θέσεις. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Σύνοδο της Ολομέλειας. Θα ήθελα καταρχήν να σας ε, κοινοποιήσω δύο λυπηρές πληροφορίες. Χθες στη, Φλωρέδη, στη Φλωρεντία κάποιος ε, πυροβόλησε δύο ανθρώπους ε, για ρατσιστικούς λόγους και για μια ακόμη φορά έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι που ήθελαν να ζήσουν και να εργαστούν στην Ευρώπη. Αυτό είναι εξαιρετικά λυπηρό και σίγουρα θα πρέπει αποφασιστικά να μην φυστούμε προσπαθειών και να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε ε, δραστηριότητα ρατσιστική, ξενοφοβική. Ε, εξίσου θλιβερή είδηση είχαμε και από το Βέλγιο, γιατί είχαμε μια τραγωδία στη Λιέγη που έπληξε αθώους ε, ανθρώπους.